Please, colleagues. Sorry, colleague. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Please take place so we can start. It's 10 o'clock. Καθίστε παρακαλώ γιατί είναι 10 η ώρα. Ας ξεκινήσουμε. Ε, περασμένες 10 για την ακρίβεια. We can start with the first part. Θα αρχίσουμε με το πρώτο τμήμα. Allora, ε, iniziamo ε, i lavori di questa seduta di commissione. 9 με 10 έγινε η συνεδρίαση των συντονιστών. Συνεχίζουμε με την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής. Α δούμε πρώτα τα τυπικά σημεία τη ημερήσια διάταξη και μετά θα σα ενημερώσω για του συντονιστέ. Καταρχήν, έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξή μα προβλέπει η συζήτηση τη έκθεση Βαλεάν για την ηθαγένεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 με εισηγητή τον κύριο Σαλαβράκο μία συζήτηση για και των εκθέσεων για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο και το Βουκουρέστι και ε, διάφορες αναφορές για πυρηνικά εργοστάσια, για τα οποία φυσικά θα γίνει συζήτηση. Οι συνάδελφοι Έφνερ και Ντεμπρούν μας ε, ενημέρωσαν ε, για την απουσία τους ε, από τη σημερινή συνεδρίαση για λόγους υγείας και ο κύριος Μπούλαντ επισκολίεται λόγω προβλημάτων συγκοινωνιών. Θα έρθει με καθυστέρηση κατά τις 11 παρά 20, ε, παρά 20 11 παρά 4 Έστειλε όμω γραπτό παρατηρήσει του, ε, θα στείλει γραπτό παρατηρήσει του για την έκθεση Βαλεάν. Ο κύριο Ιτουργκάη πρότεινε αναβολή του σημείου 18. Οπότε ακυρώνεται το σημείο 18. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Βαλεάν έχει οριστεί η διορία ε, για την κατάθεση τροπολογιών στις 19 Ιανουαρίου και την επόμενη Τρίτη στο Στρασβούργο θα συνεδριάσει ο εισηγητής με τους και εισηγητές. Σε ό,τι αφορά τις ε, αναφορές που έχουμε στη σημερινή σε διάταξη, θα παραστούν αναφερόμενοι το σημείο 12, 13, 14 και 15. 7, αυτοί θα είναι οι παρόντες αναφερόμενοι. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντίρρησεις, ε, μπορούμε να οριστικοποιήσουμε και να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ας εγκρίνουμε τώρα και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 21ης και 22ης Νοεμβρίου. Δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπω αντιρρήσεις, ε, στάσεις, οπότε εγκρίνονται και τα πρακτικά της συνεδρίασης 21ης και 22ης Νοεμβρίου. Να σας υπενθυμίσω, συναδελφοί, ότι η συντακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στις 23 Ιανουαρίου στις 4.30 το απόγευμα. Και μάλιστα υπάρχει παράρτημα το του φίλου της Προεδρίας που σας εστάλει πριν από μία εβδομάδα και ζητάτε νέο άνοιγμα της αναφοράς 803 του 2006. Έχει όμως υποβληθεί ένσταση από τον κύριο Τουργκάης ό,τι αφορά το νέο άνοιγμα αυτής της αναφοράς. Ο κύριος Τουργκάης ισχυρίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του αναφερόμενου που υπευλήθη πριν από μερικές εβδομάδες. Για το θέμα αυτό έγινε συζήτηση και τη συνεδρίαση των συντονιστών μας, την πρωινή. Θα σας ενημερώσω για τα συμπεράσματα των συντονιστών αργότερα. Και η τελευταία ανακοίνωση της Προέδρου αφορά ένα θέμα που σας έχει διανεμηθεί μία έκθεση της ΣΤΟΑ με θέμα το σύστημα των συστημάτων πληροφορικής για την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Πρόκειται για ενδιαφέρον έγγραφο, σας έχει μοιραστεί προς ενημέρωση κρίναμε σκόπιμο να σας το στείλουμε για να το διαβάσετε και ενδεχομένως να υποβάλλετε και εσείς κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση του έργου της Επιτροπής και την καλύτερη προαγωγή της ε, συμμετοχής των πολιτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών, Είχαμε στο πρόγραμμα της ε, αποφάσεις για την ανάθεση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων. Οι συντονιστές συμφώνησαν ε, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2011 να δοθεί στην ομάδα των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, ECR. Η γνωμοδότηση για τα προγράμματα ε, για την ηθαγένεια ε, στην ΑΛΔΕ και οι υπόλοιπες τρεις γνωμοδοτήσεις και κυρίως ε, η έκθεση για την εφαρμογή της εφαρμογής, έπρεπε εφαρμογής του κοινωτικού δικαίου ή της συμμετοχής των πολιτών στις επιχειρήσεις της ΣΑΜΚΟ ή την, την οδηγία πλαίσιο για το είδωρα αρμόδια καθήλια Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, είπαμε ότι για τις τρεις αυτές γνωμοδοτήσεις θα εφαρμοστεί η μέθοδος DONT και με βάση αυτή την μέθοδο θα δούμε ποιες ε, ομάδες έχουν σειρά για να αναλάβουν αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τους πολίτες, την πρωτοβουλία των πολιτών, ενημέρωσα τους συντονιστές για την πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής ΑΦΚΟ, του κ. Κασίνη, για να συμμετέχουμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής στις 26 Ιανουαρίου. Στις 26 Ιανουαρίου θα γίνει στην Επιτροπή ΑΦΚΟ η συζήτηση της έκθεσης Γκουρμάη, που αφορά τον κανονισμό για την πρόταση της πρωτοβουλίας των πολιτών. Εμείς ε, με συμφωνία όλων των ομάδων, έχουμε καταθέσει τροπολογίες προς την έκθεση Γκουρμάη με υπογραφή της Προέδρου για να βελτιώσουμε την έκθεση Γκουρμάη. Οπότε, ανοιχτή πρόσκληση, όποιος το επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος στη συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου της Επιτροπής ΑΦΚΟ προκειμένου να ενισχυθεί η πρόταση της Επιτροπής Αναφορών και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών ε, και την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής ΑΦΚΟ έχουν μερικέ φορές ε, αντίθετε απόψει από εμά, οπότε όσο περισσότεροι βρεθούμε στην συνεδρία της Επιτροπής ΑΦΚΟ, τόσο πιο ενισχυμένη θα παρουσιαστεί η δική μας θέση. Ο κύριος Μποστινάρου πρότεινε να συμμετέχουν στην συνεδρίαση αυτή όλοι οι συντονιστές της ε, Επιτροπής Αναφορών και ή δυνατόν και οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η τεχνική ομάδα εργασίας που έχουμε συγκροτήσει για το θέμα αυτό. Θα συνεδριάσει στις 17 του μήνα στο Στρασβούργο για να γίνει μια προετοιμασία για τη συζήτηση στην ΑΦΚΟ. Έχει μοιραστεί και από την γραμματεία ένα συγκεφαλαιωτικό έγγραφο, μια γενική επισκόπηση της παρουσίας των αναφερομένων πέρυσι, καθώς και το κόστος της επιστροφής των ταξιδιωτικών εξόδων. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες και δείχνουν πώς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Επισμάθηκε η ανάγκη να βελτιώσουμε τους χρόνους, να επισπεύσουμε τους χρόνους ό,τι αφορά την ε, προφορική ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών, να επισπεύσουμε τις εργασίες και να καταθέσουμε το συντομότερο δυνατόν στην Ολομέλεια αυτή την προφορική ερώτηση. Δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη σε συγκεκριμένη Ολομέλεια, αλλά υπάρχει επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί το συντομότερο δυνατόν. Άλλωστε, θα εξεταστεί όσον ούπο και η οδηγία για, τις, ε, για τους αναπήρους. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να εξετάσουμε το συντομότερο δυνατό αυτή την προφορική ερώτηση για τους τυφλούς. Ως πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Αναφορών θα ζητήσω από το Προεδρείο να επισπεύσει τη συμπερίληψη της προφορικής αυτής ερώτησης στην σε διάταξη της Ολομέλειας. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις, οπότε αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για την έκβαση της συνεδρίας των συντονιστών θα έλεγα να περάσουμε στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της τακτικής μας συνεδρίασης που είναι το σημείο 7 και προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης Βαλεάν στην οποία θα δώσω και το λόγο για να μας κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, για την έκθεση σε ό,τι αφορά την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρση των εμποδιών στα δικαιώματα των πολιτών, άκουσα πολύ προσεκτικά όλες τις προτάσεις και όλα τα σχόλια και προσπάθησα να τα συμπεριλάβω στο σώμα της έκθεσής μου. Εξού και θα επικεντρωθώ στην παρουσίασή μου στα κυριότερα ζητήματα τα οποία μου ετέθησαν υπόψη από τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα, υπό την ε, οπτική γωνία της οδηγίας για την ελεύθερη μετακίνηση έχουν ε, περάσει από τα χρόνια από την θέση ισχύ της οδηγίας αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της. Περισσότερες καταγγελίες έχουν να κάνουν με το δικαίωμα εισόδου, διαμονής για περίοδο άνω των τριών μηνών, ε, ε, την ισχύ των αδειών διαμονής, ε, δια, δικαιώματα επανένωση οικογενειών, μόνιμης διαμονής κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει, και αυτό ζητώ στην έκθεση, να μεταφερθούν οι διατάξει τη οδηγία για την ελεύθερη μετακίνηση ε, σωστά και να ελοπιθούν σωστά από τα κράτη-μέλη. Και αν χρειαστεί, θα πρέπει να κινήσει διαδικασίε επί παραβάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να άρουν τα πρακτικά και άλλα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και να ε, θέσουν ένα ε, τέρμα σε ε, δυσκίνητε, αδικαιολόγητες διοικητικέ διαδικασίες οι οποίες περιορίζουν την εφαρμογή αυτού του δικαιώματο. Η έννοια της ηθαγένειας γίνεται πολύπλοκη σε ό,τι αφορά τους Ρωμά, στο πλαίσιο δηλαδή ε, κάποιων απελάσεων που είδαμε και ε, στη Γαλλία το 2010. Κάτι το οποίο συνιστά παραβίαση της, αρμο... της ε, οδηγίας αλλά γίνεται κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέματα δημόσιας ασφάλειας μπορούν να τεθούν αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση ή εθνική, φιλετική καταγωγή, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την αυτόματη απέλωση η μη ε, κατοχή παρκών οικονομικών πόρων. Θα πρέπει να λάβουμε κοινή ευθύνη για να προωθήσουμε την ένταξη των Ρωμά και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί και η διατάξη του ψήφισματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 9η Μαρτίου 2011 και οι στρατηγικέ ε, για την ένταξη μέχρι το 2020. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι η έλλειψη αμοιβαία αναγνώριση σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση ε, ζευγαριών ε, ομοφύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ελεύθερη διακίνηση όλων των πολιτών και των οικογένειών τους χωρίς διάκριση λόγω γενετήσου προσανατολισμού ή εθνικότητας. Η έκθεση επαναλαμβάνει την έκκληση προς τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τα δικαιώματα τα οποία εκχωρούνται από τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας ελεύθερης διακίνησης, όχι μόνο ε, στα ομοφυλά ζευγάρια, αλλά και όταν υπάρχει σταθερή ε, σχέση, ακόμη και αν είναι ομόφυλα τα ζευγάρια με βάση την αναγνώριση, ε, ε σεβασμό της αξιοπρέπειας, ε, σεβασμό της ιδιωτικής, της προσωπικής ζωής. Χαιρετίζουμε επίσης την πρώτη της έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκή Ένωσης, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα μπορούν λοιπόν ε, οι πολίτες να βασίζονται ε, στο χάρτη αυτό και στα δικαιώματα αυτά. Αλλά με ανησυχεί το γεγονός ότι η πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαίου Μεσολαβητή ε, κατέληξε στο ότι τα 72% των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι παρκώς ενήμεροι για το χάρτη. Ζητούμε λοιπόν από την Κομισιόν στο μέλλον να επικεντρωθεί όχι μόνο στην εφαρμογή του χάρτη, αλλά και σε όλα τα άρθρα τη Σύνδεξη Ευρωπαϊκή Ένωση που σχετίζονται με θεμελιώδη δικαιώματα, κατάσταση θεμελιών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να εξηγήσει, να προωθήσει καλύτερα η Κομισιόν όλες αυτές τις μεριώδεις διατάξεις. Επίσης, συμπεριέλαβα στην έκθεση κάποιες παραγράφους οι οποίες έχουν να κάνουν με το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα. Διότι φυσικά και είναι καλύτερο να υπάρχει στον δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο διαφανή. Επίση, ε, να μπορούν να δοθούν κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά την έρευνα από την Κομισιόν χωρίς να ανατίθεται, να υπονομεύεται η ίδια η έρευνα και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε φακέλους αυτούς, ιδίως όταν μιλάμε για ε, προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας ε, υγείας και υπάρχει κίνδυνος μια βλάβη, η ζημία έτο 2013, έτο Ευρωπαίων πολιτών. 20 ε, χρόνια δηλαδή από την εισαγωγή της έννοιας της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Αυτό σίγουρα δεν είναι ένα σημαντικό έτος. Θα πρέπει να γίνουν πιο γνωστά τα δικαιώματα ε, που συνεπάγεται η έννοια αυτή και θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες ε, για την πρόθεση των δικαιωμάτων των πολιτών. Όπω είπε και η πρόεδρος, να σας υπενθυμίσω και εγώ την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση ή τη 19 Ιανουαρίου. Προς το παρόν, αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαλέαν για την παρέμβαση, την έκθεση. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βαλεάν, τη συνάδελφο, για την έκθεση. Και πιστεύω ότι η συζήτηση για την έκθεση είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο των συζητήσεων για την κινητικότητα των Βουλγαρών και Ρουμάνων πολιτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ήθελα να επισημάνω το σημείο 8 της εκθέσεως Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από τα κράτη-μέλη ε, με έγγραφά του την αξιολόγηση της κατάστασης. Η έκθεση κυρίας Βαλεάν ακολουθεί τις επιλογές Μαρινέσκου και Βαλεάνου του Δεκεμβρίου του 2011 και θα ήθελα να επισημάνω την ε, ανάγκη για περίληψη των ΡΟΜ μέσα στην εθνική στρατηγική. Όπως καταγράφεται αρρώστη και στην παράγραφο των Ρωμά, την ε, παράγραφο 12. Στο τέλος του 2011 υπευλήθη πρόγραμμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ σκοπεύω να καταθέσω προτάσεις ε, για να ε, στηρίξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες στα δικαιώματά τους. Θα ήθελα εδώ να πω ότι ε, έχουμε εξελίξει το τομέα αυτόν, θα πρέπει να τις καταγράψουμε. Ήθελα να υποστηρίξω την έκθεση και την κυρία Βαλέων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπέκερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τη συνάδελφο για την έκθεση αυτή όντως είναι μια πολύ χρήσιμη βάση για τις εργασίες μας. Και θα ήθελα να συμπληρώσω με τις εξής ε, παρατηρήσεις, ξεκινώντας όμως, όμως με μια συγγνώμη, διότι δεν ε, υπέβαλα τις προτάσεις μου εγκαίρως στην κυρία Βαρεάν, θα το πράξω στο εγγύς μέλλον, ε, στο συγνώμη που δεν έδωσα τις προτάσεις αυτές εγκαίρως, νωρίτερα. Ξέρετε ότι με απασχολούν πολύ τα θέματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το γενικότερο θέμα της πρόσβασης και της κινητικότητας ξεκινάει με δεδομένα τα εμπόδια στην κινητικότητα, από αυτά ξεκινάει, ε, τα επεκτείνει την εξέτασή του η κυρία Βαλέαν, τα αναλύει και κάνει προτάσεις, τις οποίες ε, συμμερίζομαι και εγώ. Ωστόσο πιστεύω ότι καλό θα ήταν να ε, καταγραφούν πιο ξεκάθαρα κάποιες προτεραιότητες μέσα στην έκθεση και δει εκείνες οι οποίες Ε, υπογραμμίζουν την έννοια ότι είναι πολύ λίγες οι γνώσεις που έχουν οι πολίτες για το τι σημαίνει το να ζει κανείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα εμπόδια ε, αποδιαρθρώνονται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί μη τι άλλο σε κάποιο είδου προήμιο τη εκθέσεω, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτού του στόχου. Βεβαίως, δηλαδή θα πρέπει να δοθεί ε, έμφαση στην ιδέα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης του πολίτη. Όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, κάποιο πρόσκομα, να γνωρίζει τι δυνατότητες έχει και τι δικαιώματα. Σε αυτό νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να αποδεχθούν αυτά τα προσκόμματα. Επίσης, και πιστεύω ότι χρειάζεται να αναλυθεί η δράση στον εξή τομέα, ότι η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά και ανθρώπους οι οποίοι δεν κινούνται εκτός των συνόρων της χώρας τους, αλλά αναλαμβάνουν δραστηριότητες υπερσυνοριακές. Φερρυπίν, μια ε, κληρονομιά πέραν των συνόρων ή διαδικτυακές αγορές, αγοραπολισίες. Αυτά είναι άλλες δραστηριότητες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κινητικότητα των πολιτών και θα ήθελα πολύ πιο επακριβείς ορισμούς, γιατί εάν κοιτάξουμε και την έκθεση Κόσερε παραδείγματι, εκεί που γίνεται λόγος για ανθρώπους με αναπηρία, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένε πτυχές, εξειδικευμένες αν θέλετε, οι οποίες μπορεί να αφορούν μόνο άτομα με αναπηρία, αλλά θα ήθελα και αυτό να το λάβουμε υπόψη και να παραπέμψουμε ενδεχομένω την έκθεση αυτή. Αν μου επιτρέψετε λοιπόν, θα ήθελα να σας υποβάλω τις σχετικές προτάσεις, έστω μια μικρή καθυστέρηση, για να γίνει σχετική συμπλήρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ζανόκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω ο, την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου για την έκθεση. Ιδιαίτερα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε συνάδελφος. Και θα ήθελα να ξεκινήσω μια ερώτηση. Ξέρουμε ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει και την αντίστοιχη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010. Στο σημείο 24 λοιπόν λέτε ότι προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στη σύνταξη νέα έκθεση για την Ιθαγένεια του 2013. Αν δεν είναι καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτό, αφού το έτος ηθαγένειας είναι το 2013. Δεν θα έπρεπε η έκθεση να είναι διαθέσιμη πριν από την άνοιξη του έτους ηθαγένειας. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να αναλογιστούμε και σε ποιο βαθμό η Επιτροπή ε, δραστηριοποιείται στην εκδοση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και τα δικαιώματά του. Και θα ήθελα επισήμω να διατυπώσω ανησυχία, διότι βλέπω ότι πολλά ακόμα υπολείπονται να γίνουν. Εγώ έχω συντάξει γνωμοδότηση εκ μέρου τη Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών για την ίδια αυτή έκθεση. Και πρέπει να πω Μάλιστα είχα μία σελίδα προτάσεων με πέντε θέσεις και σε αυτή τη μία σελίδα έλαβα 74 τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την γνωμοδότηση στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών στις 25 Ιανουαρίου και ελπίζω η Επιτροπή των Αναφορών να μπορέσει να αξιοποιήσει τις συστάσεις μας. σε ορισμένα και πολύ ευαίσθητα ζητήματα ίσως να υπάρξουν, ε, ίσως να διαπιστωθεί απόκληση απόψεων. στο κατά πόσον θα χορηγούνται πλήρη δικαιώματα ως προς την επανένωση των οικογενειών, οι ε, ομοφιλόφιλες οικογένειες, τέτοια ζητήματα. Επίσης, κάποιες πολιτικές ομάδες αντιτάσσονται στην ε, ιδέα για προσφυγή κατά κράτους μέλους σε παραβάση όταν δεν τηρούν αυτά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες. Η κυρία Βαλεάννα ήδη επεσήμανε το πρόβλημα των Ρωμά στη Γαλλία και κύριες διαφωνίες που αναδύονται μεταξύ των πολιτικών ομάδων έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των δικαιωμάτων μονίμου κατοίκου στους ε, υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων κρατών δηλαδή αφετέρου. πολιτική μου ομάδα και θα ήθελα να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου ε, προς άλλες πολιτικές ομάδες και μέλη τους που με υποστήριξαν, προτείνει μία φόρμουλα που θα έλεγε ότι τα δικαιώματα των μόνιμων ε, κατοίκων μπορούν να πλησιάσουν τα δικαιώματα, μπορούν να μοιάζουν με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηθαγένειας δηλαδή. Ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει και νωρίτερα με την Επιτροπή των ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Την έκθεση αντίστοιχα είχε κάνει και η Επιτροπή των Αναφορών στο παρελθόν. Είχαμε την έκθεση Λάζιξ το 2009. Αυτά λοιπόν. Και ελπίζω οι προτάσεις μας όπως θα προκύψουν με την ψηφοφορία της 25ης Ιανουαρίου στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, να αξιοποιηθούν και να ενσωματωθούν στην έκθεση της Επιτροπής των Αναφορών. Και όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε να οδηγήσει σε περαιτέρω και θετικές εξελίξεις στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Βαλεάν για την έκθεσή της και να τη διαβεβαιώσω για την αμέριστη υποστήριξη της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Επίσης, ε, θα ήθελα να εξάρω το πολύ πλούσιο περιεχόμενο αυτής της έκθεσης που βρήθη ιδεών και που μιλάει για την έμπρακτη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου προκειμένου να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και να μειωθεί η απόσταση μεταξύ του θεωρητικού χαρακτήρα των κοινοτικών εγγράφων και τις ε, πρακτικές πτυχές καθημερινότητας των πολιτών. Γιατί εκεί είναι που πονάει η καθημερινότητα και τα προβλήματά της. Και ως προς αυτό, ως προς τη μείωση αυτής της απόστασης μεταξύ θεωρίας και πράξης, η έκθεση είναι πολύ σημαντική. Σε αυτό το πλαίσιο της ε, οικονομικής κρίσης και της διάσωσης της Ευρωζώνης είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για την οικονομική διακυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό να μην ξεχνάμε και την άσκηση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στην καθημερινότητά τους. Διαφορετικά ε, θα κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε με μία ε, απόμακρη και ψυχρή Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που θα πληρώσουμε σε επόμενες ευρωεκλογέ αν οι πολίτες απομακρυνθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καλό θα ήταν επίσης να φροντίσουμε για να έρθουν όλα τα εμπόδια που επισημαίνει η κυρία Βαλεάν. Να κάνουμε έναν απολογισμό, μια απογραφή όλων αυτών των δυσκολιών και των εμποδίων από την Επιτροπή. Να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση, την άρση αυτών των εμποδίων για να ε, ενισχύσουμε το ρόλο μας, ε, ρόλο προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν κάποια δημοκρατικά και θεμελιώδη δικαιώματα που ασκούνται ε, από τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, καταστρατηγίες τέτοιων δικαιωμάτων που παρατηρούνται στην Ουγγαρία σε ένα κράτος μέλος. Και καλό θα ήταν να επισημάνουμε εδώ το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής μας στην προσπάθεια προάσπισης των δημοκρατικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Θα ήθελα εν τέλει να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Βαλεάν για την έκθεσή της και να πω στην Πρόεδρο την κυρία Ματζόνη που μας υπέβαλε ε, στατιστικές ε,